Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε με το σημείο 1. Η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Με τα ακόλουθα σχόλια. Σημείο 13. Έχουμε την πρόταση για συγχώνευση μεταξύ της ΕΠΟΛ και της Να βάλετε το σημείο αυτό. Ο κύριος Μπάφη δεν μπορεί να παρευρεθεί και έχουμε και το σημείο 14 για την αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προχωρούμε. Στο σημείο 3, η κατάσταση των συνεχιζόμενων διοργανικών διαπραγματεύσεων στις νομοθετικές διαδικασίες, αλλά η κυρία Αντωνέσκου δεν είναι εδώ. Uh, Δεν είναι εδώ σήμερα το πρωί. Πρόκειται για την πρόταση οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Και θέλω να σας ενημερώσω για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, απουσία της εισηγητρίας. Τελευταίος τριμερής διάλογος, ο έκτος, έλαβε χώρα χθες το απόγευμα. Το αποτέλεσμα θα θεωρηθεί θετικό, έγινε πρόοδος και οι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που ήταν ιδιαίτερα αποκλίνουσε στην αρχή σιγά σιγά έρχονται πιο κοντά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία το Κοινοβούλιο όπως η αρχή του απορρίτου στις επικοινωνίες, στην επικοινωνία μεταξύ του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και του δικηγόρου η Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή της να παραπέμψει το θέμα στην Κορεπέρ στις 27 Μαρτίου και οι παρεκκλήσεις ε, στο άσκηση των δικαιωμάτων που υπάρχουν στην οδηγία, προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων και πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση για άτομα που υπόκειται στο Ευρωπαϊκό Έντερμα είναι ακόμη ανοιχτά. Η που σκοπεύει να συνεχίσει σε στενή συνεργασία με τους Κιώδης προκειμένου να φτάσει σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης των κισμέλων. Επόμενος τριμερής διάλογος ε, θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στο Στρασβούργο και ίσως ένα ακόμη το Μάιο. Αφού ακούσατε λοιπόν ε, πώς έχει η κατάσταση, η για το φάκελο αυτό, προχωρήσουμε στο σημείο 4 το οποίο έχει να κάνει με τα κύρια έγγραφα για τα κύρια επενδυτικά προϊόντα. Ο κύριος Δίας Δεμέρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Πάτε πολύ γρήγορα σήμερα το πρωί, δεν διαφωνώ, ίσως εγώ να πηγαίνω αργά. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω ένα λεπτό στο σημείο 3 που έχει να κάνει με την εξέλιξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Απλώς για να κάνω μια μικρή δήλωση. Μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να μιλήσω για τις κατεξουσίες πράξεις, για τις εκτελεστικές πράξεις του μαθητική διαδικασία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σκέψη. Ήδη ξέρουμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν σε σχέση με τις καθεξουσιοδότηση πράξεις και επίσης γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αδιαφεσβήτητα. Αντίθετα, το Συμβούλιο παραμένει σε μια θέση απροσδιόριστη. Μερικές φορές λέει ναι, μερικές φορές όχι. κάτι που έχει να κάνει με την τροποποίηση του κανονισμού 539-2001 θα προτείνουμε να ψηφιστεί στην Επιτροπή στις 8 Απριλίου. Στο φάκελο αυτό θα διατηρήσουμε την ε, επιλογή των ε, της πράξεων για δύο θέματα, για την αναστολή και για την εμβαιότητα. Με ποια πρόθεση, με την πρόθεση να διατηρήσουμε ενοποιημένη και ξεκάθαρη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα να εξαναγκάσουμε σε ισχυρές διαπραγματεύσεις από την στιγμή που θα ακολουθήσει αυτή την ψηφοφορία μέχρι αυτή η ψηφοφορία να πάει στο Κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, μετά από τη δήλωση που μόλις έκανα, θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια προσέγγιση σε σχέση με τη χρήση εξουσιοδότηση πράξεων μεταξύ των τριών οργάνων, αν υπάρχει κάποια τέτοια προσέγγιση. Πρόεδρος, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Εμείς σημειώνουμε το όσα μας είπατε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να συνεχίσουμε αυτό το χάρτη πορεία σε σχέση με το φάκελο 539 του κανονισμού 539-2001. Και απλώς να σχολιάσω ότι η προβληματική σχέσεις Κοινοβουλίου Κομισιών σε σχέση με τις κατεξουσιδότητες πράξεις συζητήθηκε εκτενώς στην τελευταία συνεδρίαση των Προέδρων των Επιτροπών στην διάσκεψη των Προέδρων, των, προέδρων, των Επιτροπών. Άτυπη διάσκεψη των Προέδρων ήταν αυτή. Έτσι ώστε ε, οι Πρόεδροι ε, να προβληματιστούν επί του θέματος αυτού μια συγκεκριμένη μέρα που ορίζεται για αυτό το ζήτημα αν ε, αυτή η προβληματική παρουσιάζεται έντονα και σε άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος ή Μεταφορών, ε, ναι, να είναι έντονη και αυτή η προβληματική, αλλά όχι τόσο εδώ. Βέβαια, εμείς το σημειώνουμε. Να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε συνεδρία συντονιστών. Στις 11.30 νομίζω προβλέπετε. Έχουμε κάπως ε, περίεργη μέρα σήμερα. Και στις 6.30 ε, και κλεισμένο το θερμό θα έχουμε μια συζήτηση με την Επίτροπο Μάλστρομ ε, για τα θέματα Σέγγεν και την επιπλοκή τους. Όμως στις 11.30 συντονιστές θα συζητήσουμε το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. και συγκεκριμένα τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους φακέλους που υπάρχουν σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Το σημειώνουμε και μετά τη συνεδρία των συντονιστών η συντονίστρια του ΕΛΚΑ, η κυρία Ματιέ, θα μπορέσει να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της συζήτησης αυτού του σημείου στις συνεδρίες των συντονιστών. Κύριε Μέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ε, θετική ανταπόκρισή σας στο έτοιμά μου. Μάλιστα, αφού τα σημειώσαμε αυτά, λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε τώρα να ξαναπάμε στο σημείο 4, το οποίο το είχα ανακοινώσει και έχει να κάνει με τα κύρια έγγραφα πληροφόρησης σχετικά με τα μελλοντικά προϊόντα. συγκητής είναι ο συνάδελφος Πέτρου Κωνσταντής Λούχαν. Βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Απλώς να πω ότι στις συνεδρίες της 21ης Φεβρουαρίου ο κύριος Λούχαν παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησης για αυτή την πρόταση κανονισμού. Η ημερομηνία για την κατάσταση τροπολογιών είχε οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου. 35 τροπολογίες κατατέθηκαν. Και μαζί με αυτές που παρουσιάστηκαν από τον εισηγητή φτάνουμε στις 48. Επομένως, μετά από τη συζήτηση αυτή που θα έχουμε σήμερα, στην οποία θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, η ψηφοφορία θα μπορούσε να λάβει χώρα στις 8 Απριλίου, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Να ακούσουμε τώρα τον εισηγητή. Και κατόπιν μπορούμε να ακούσουμε και εκπροσώπους Κομισιόν και Συμβουλίου. Παρακαλώ. Κύριε Λούχαν, έχετε το λόγο. Muchas gracias, señor presidente. It's a quite technical report actually. We had to provide a... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν τεχνικό το ζήτημα επί του οποίου κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε. Αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για βασικά ε, ε, έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα. Ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά και πάλι επειδή σχετίζεται με πολλά θεμελιώδη δικαιώματα το θέμα, κρίθηκε απαραίτητο να γνωμοδοτήσει και δική μας Επιτροπή. Η πρόταση σκοπό έχει να βελτιώσει τη διαφάνεια στην αγορά επενδύσεων για τους μικροεπενδυτές. Τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές έχουν καταστεί πάρα πολύ δύσκολα και δυσνόητα και γι' αυτό οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν απαραίτητα να τα αξιολογήσουν και να τα συγκρίνουν τα προϊόντα αυτά γιατί υπάρχει ασυμμετρία πληροφοριών. Αυτή η πρόταση λοιπόν θέτει πιο σαφείς κανόνες και υποχρεώσεις για τα χρηματοοικονομικά πιστοτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν στον επενδυτή για να βελτιωθεί η κατανόηση των προϊόντων και να είναι και πιο εύκολη η σύγκρισή τους. Επίσης, δίνει μεγαλύτερη δύναμη στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβιάσεις ενδεχόμενες των υποχρεώσεων των οργάνων αυτών. Όπως σας είπα, η Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι η αρμόδια Επιτροπή. Εμείς κληθήκαμε να εξετάσουμε τεχνικές πτυχές για να υπάρξει άμεση σύνδεση με τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μιλάμε ιδιαίτερα για επενδυτικά κεφάλαια με προϊόντα για τους μικροεπενδυτές και κάποιες, ε, κάποιου είδους ε, ε, ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς. Όπως είπατε, έχουν κατατεθεί 48 τροπολογίες δεν έχουν να κάνουν όλες ε, με το κάθε αυτό αντικείμενο της ΛΥΜΠΕ, αλλά έγιναν αποδεκτές, γίνονται αποδεκτές επειδή έχουν να κάνουν με την έκθεση προφανώς. Ιδιαίτερα η κυρία Βάιντεν Χόλτζερ κατέθεσε πολλές τροπολογίες. Όπως σας είπα, δεν ε, σχετίζονται όλες απαραίτητα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, πολλές τροπολογίες θα αυξήσουν την διαφάνεια για τον καταναλωτή, για τον ιδιώτη. Θα γίνει κατηδίαν συζήτηση με την κυρία Βάιντεν Χόλτσερ για να κάνουμε κάποιες εμβιβαστικές προτάσεις τελικά. Η συζήτηση θα ξεκινήσει σήμερα. Ο κύριος Ταβάρης επίσης κατέθεσε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Έχουμε ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο εξέβρεση συμβαστικών προτάσεων με το γραφείο του. Και όπως είπατε, στις 8 Απριλίου θα ψηφιστεί η έκθεση. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει και η Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Λούχαν. Τώρα καμιά συζητησούλα. Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Είδα όμως και τον κύριο Μπρόγκς που ζήτησε το λόγο, τίποτε κανείς άλλος. Κύριε Μπρόγκς πρώτος και καλύτερος. Ναι. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτό που άκουσα είναι η θετική. Προφανώς χρειάζονται προστασία αυτά τα επενδυτικά προϊόντα για να γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Προτιμώ φυσικά τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα προστατευτικά μέτρα γιατί εκεί να γνωρίζουν καλύτερα <clears throat> τις ανάγκες. Ας το αφήσω όμως προς το παρόν. Ο εισηγητής μας λέει ότι θα προτιμούσε κανονισμό. Εγώ θα έλεγα αν χρειαστεί νομοθεσία καλύτερα να είναι, έχει μορφή οδηγίας που να επιτρέπει τουλάχιστον περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή της. Εκ πρώτης απόψεως φαίνεται να πρόκειται απλώς για ένα μέτρο προστασίας των καταναλωτών Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι υποτιμητικό, αλλά υπάρχει και ένας άλλος στόχος, όπως και σε άλλα μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Φαίνεται από την τέταρτη παράγραφο ότι λέει ένα ομοιόμορφο σύστημα στην Ένωση που να διευκολύνει τη σύγκριση των προϊόντων. Άρα ο κύριος στόχος είναι όχι απλώς προστασία των καταναλωτών, αλλά διευκόλυνση της ενιαίας αγοράς. Σταματάω εδώ. Βάιντεν Sie haben das Εκτός μικροφώνου. Σε ό,τι αφορά την ε, προσφορά των προϊόντων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Θεωρώ ότι είναι καθυστερημένη αλλά σωστή αντίδραση αυτή στην οικονομική κρίση και ασφαλώς θα παίξει σημαντικό ρόλο η Επιτροπή μας. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν ισχύουν μόνο για τους παρόχους αλλά και για τους μικροεπενδυτές. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινούνται οι τροπολογίες μου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θέλει να το συζητήσει ο εισηγητής. Γενικά αυτό που θεωρώ ότι είναι ε, σημαντικό είναι να περιοριστεί ο περίπλοκος χαρακτήρας των προϊόντων αυτών, γιατί για τον πολύ κόσμο είναι ακατανόητα. Και θα πρότεινα σε κάθε περίπτωση να εισαχθεί ε, μια ιδεολογική σκέψη, η οποία θα υποδεικνύει αυτή την πτυχή που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε γενικές γραμμές. Συμφωνώ με τις θέσεις του εισηγητή. Τρία σημεία θα ήθελα να κάνω κάποιες προσθήκες, κάποιες διορθώσεις σε ό,τι αφορά τη μείωση των εξαιρέσεων, γιατί προβλέπονται πάρα πολλές εξαιρέσεις στην παρούσα φάση. Οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει καταρχήν να διατίθενται για όλα τα προϊόντα. Δεν υπάρχει λόγος γιατί, για τον οποίο ε, κάποια προϊόντα θα έπρεπε να εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Επίσης το θέμα είναι και το περιεχόμενο των ε, πληροφοριών στο άρθρο 8 και αυτό κινείται προς την κατεύθυνση της χρωματότητας της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πότε μπορεί κανείς να τερματίσει σχετικές συμβάσεις ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά και να μην τίθεται και θέμα προσβασιμότητα στι πληροφορίε, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο κατάχρηση. Πραγματικά θα πρέπει να αποφευχθούν τέτοιες ε, καταχρήσει. γενικά. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό θέμα για, από άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι η, ο κατανοητός χαρακτήρας των πληροφοριών αυτών. Μόνο τότε θεωρώ ότι προστατεύονται τα τα δικαιώματα του πολίτη. Και τέλος βλέπουμε ότι ένα πρόβλημα της κρίσης ήταν και είναι η μείωση της εμπιστοσύνη του πολίτη. Θεωρώ λοιπόν ότι μειώνοντας τις πληροφορίες που παρέχονται θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε αυτή την συρρυκνούμενη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν ε, δεν θέλει άλλο το λόγο από τους συναδέλφους, για ένα λεπτό, να ακούσουμε εκπροσώπους από την Κομισιόν ή από την Προεδρία. Θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ, Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντική αυτή η συζήτηση γιατί η συζητηση γιατι την προθεση αυτής της πρότασης ε, είναι ιδιαίτερα κατανοητή. Αυτή η πρόταση εστιάζεται στην βελτίωση της κατανόησης και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών. Έχει μια πτυχή ενιαίας αγοράς, αλλά αφορά την προστασία των καταναλωτών και αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Γιατί ξέρουμε ότι το κύριο πρόβλημα στα επενδυτικά προϊόντα λιανικής είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν τα προϊόντα που τους πολλούνται και να συγκρίνουν τα προϊόντα αυτά. Έτσι λοιπόν κάποιος δεν καταλαβαίνει δεν μπορεί να συγκρίνει τα προϊόντα. Είναι δύσκολο να υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική αγορά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλαμβάνουν οι αγοραστές τι δεσμεύσεις να λαμβάνουν. Όλα αυτά συνάδουν κατά την άποψή μας και η έρευνα που κάναμε πριν την παρουσίαση της πρόθεσης αυτής υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση απέναντι έναντι διάφορων ε, προϊόντων και να χρησιμοποιούνται τα ίδια πρότυπα σε ό,τι αφορά τι ε, πληροφορίε. Δηλαδή να υπάρχουν ήδη τίτλοι για τα προϊόντα έτσι ώστε να μπορούν ε, οι πολίτες να καταλάβουν και να χρησιμοποιούν τι πληροφορίε για τη σύγκριση. Αυτή είναι μια κύρια αρχή που διέπει την πρότασή μα. Αλλά γενικά είναι πολύ ενθαρρυντική αυτή η συζήτηση εδώ νομίζω. Αυτά ήθελα να σχολιάσω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάποιος από την Προεδρία θα ήθελε το λόγο ή όχι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον να επανέλθουμε στον κύριο Λούχαν, τον συγητή. Ευχαριστώ. Ως οικονομολόγος, ε, ίσως ε, κάποιος οικονομολόγος θα είχε μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου καταρχήν ε, όσους προσκευάζουν αυτά τα προϊόντα και τις υποχρεώσεις και κατά τα λοιπά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αγοραστών. Όπως σωστά είπε η Κομισιόν, τι χρειαζόμαστε. Πρέπει να κάνουμε κάτι σε νομοθετικό επίπεδο προκειμένου να είναι πιο δυναμική και πληρής η αγορά. Αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για ένα προϊόν, τότε ο αγοραστής δεν θα έχει κίνητρα να το αγοράσει. Δηλαδή, ένα από τα όπλα αυτής της ε, έκθεσης θα ήταν ε, να καταστήσει πιο αποτελεσματική την αγορά. Αλλά όχι φυσικά να ξεχνάμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα των δύο μερών και ιδίω των πολιτών. Και αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε ο κ. Μπρόγκς, υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητες, αν θα πρέπει να μιλάμε για εθνική αρμοδιότητα ή αν θα πρέπει να έχουμε γενικώ τυποποιημένους κανονισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων σε αυτή τη λιανική αγορά και επομένως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινούς κανόνες. Ε, αυτό ήταν και το κρίσιμο σημείο συζήτηση στην περίπτωσή μα, αλλά ξεκολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αρχή τη επικουρικότητα ισχύει εδώ και πρέπει φυσικά να επιμερίσουμε τι αρμοδιότητε στο επίπεδο αυτό. Αλλά θα ήταν ε, καλύτερο, θα υπήρχε πλέον έκτημα αν περισσότερες αρμοδιότητε ενέπιπταν έπιπταν στους τη της Ευρωπαϊκής σε σχέση με τη μείωση των εξαιρέσεων. Θέξατε αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης γενικά ή να δίνουμε όσο δυνατόν λιγότερες πληροφορίες ε, προκειμένου ο αγοραστής να τις θυμάται όλες αφενός, αλλά από την άλλη οι πληροφορίε αυτές να είναι και τόσο πλήρε, έτσι ώστε να γίνεται μία ορθή σύγκριση. Είμαι ανοιχτό στο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Όμω εμένα δεν μου αρέσουν οι εξαιρέσει καθόλου. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα πρέπει να σεβαστούμε τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω επειδή οι αγορέ μεταξύ των διάφορων χωρών ε, διαφέρουν και υπάρχει και ο πειρασμός και μεγαλύτερη ανάγκη και περισσότερες απαιτήσει στην αγορά να μπούμε σε νέες αγορές, ε, παραδείγματος χάρη στα κρατημέλη. Για θέματα προσβασιμότητας, προκειμένου και το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει η πρόσβαση να είναι πιο γρήγορη και πιο σωστή και πιο κεντρική. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο κόσμος και ιδιαιτέρως οι καταναλωτές έχουν επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες σήμερα και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο υπολειτουργεί κάπως το σύστημα σε σχέση με το επίπεδο που θα μπορούσε να λειτουργεί. Άρα, εμείς θέλουμε να δώσουμε μία όθηση. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, αλλά ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, τους αγοραστές των προϊόντων αυτών. Δεν είναι εύκολο αυτό, δεν πουλάμε άλλωστε φρούτα, μήλα, αχλάδια. Ο όγκος των πληροφοριών είναι ασφαλώς πολύ μεγαλύτερος από ότι στα κανονικά εμπορικά προϊόντα. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει επακριβώς να εξετάσουμε το πόσο μπορούμε να απλοποιήσουμε τις περίπλοκες αυτές πληροφορίε. πληροφορίες. Όχι όμως απαραίτητα να τις περιορίσουμε. Δεν είμαι υπέρ της μείωσης των πληροφοριών. Να τις απλοποιήσουμε, ναι. Να τις περιορίσουμε, όχι. Αυτό θα πρέπει να το ισορροπήσουμε. Τελευταίο στοιχείο, το στοιχείο της κρίσης. Ασφαλώς θα πρέπει να τεθεί στο σωστό πλαίσιο η πρόταση. Η κρίση ασφαλώς επηρέασε πολύ την αγορά των επενδυτικών προϊόντων. Και τώρα τα θεσμικά όργανα καλούνται να βρουν και αυτά έναν τρόπο εισαγωγής μέτρων ενίσχυσης, προκειμένου ο κόσμος να εξετάσει και πάλι τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να δοθεί οικονομικό κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτή είναι η άποψή μου σε σχέση με τις τρεις τροπολογίες που καταθέσατε και προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Λούχαν, τώρα Οι 48 τροπολογίες θα εξεταστούν αφού ακούσαμε την άποψη του εισηγητή και των ε, συναδέλφων. Αλλά να σας πω ότι στο σημείο αυτό Η ημερομηνία που έχει προβλεφτεί για, για την ε, ψηφοφορία είναι η 8η Απριλίου. Εδώ στην Επιτροπή εννοώ. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία που προβλέπετε για τις 10 και 4. Η ώρα είναι 10 και 5 και επειδή ξέρετε πολλοί βουλευτές έχουν προβλέψει να έρθουν στις 10 και 4 ακριβώς θα σας πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. 10 και 4 ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμφωνία για τη Μολδαβία. 10 λεπτά διάλειμμα.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

Με τις κάρτες παρακαλώ. Ε. τσακ τσακ Μάρι. Τι είναι ο επίσκοπος. Mm. Okay. If I may have your attention. Προσέξτε παρακαλώ. Καθίστε. Και εσείς κύριε Λούχαν. Κύριε Λούχαν μου. Καθίστε. Είναι 10 και τέταρτο. και υπάρχει η απαρτία. Λοιπόν, το σημείο 5. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο σύστασης για την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Μολδαβίας για τις θεωρήσεις. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι μόνο μία ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν. Αρχίζει. Τώρα έλξε όμως. Πάει. Έλξε. Έλξε. Λοιπόν, I mean, those, Αυτοί που μόλις μπήκαν να να μας πούν τι θα ψήφιζαν κυρία Γαβριήλ μία ψήφος υπέρ και η κυρία Ρομέρου επίσης. Α, και ο κύριος Έντσο. 41 υπέρ 2 κατά. Πώς? 42 υπέρ, 42 υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί τον Απρίλιο. Ευχαριστούμε. Το επόμενο σημείο τώρα. Αυτά, τελείωσε η ψηφοφορία. Τελείωσε η ψηφοφορία είπα. Τώρα, τώρα λέγω, το επόμενο, το 6. τροποποιούμε κανονισμό για τους, τις πρόδρομες ουσίες των ναρικοτικών. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Hello. <laughs> So, now, moving to point number which is... Είπα το 6. Τροποποίηση του κανονισμού για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών. Εισηγήτρια κυρία Άννα Χέντ. Έχουν κατατεθεί 25 τροπολογίες, συν τις 21 που υπήρχαν προηγουμένως, και θα συζητηθούν σήμερα, αφού μας μιλήσει η κυρία Χέντ, εισηγήτρια που έχει και το λόγο. Ευχαριστώ. Και τους συντάκτες των τροπολογιών. Όπως έχω ξαναπεί, το θέμα φαίνεται πολύ τεχνικό, αλλά είναι σημαντικό. Όσο για τις τροπολογίες, τις δέχομαι σχεδόν όλες. Οι περισσότερες αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Από την ΚΟΕ πρότειναν σχεδόν τη διαγραφή των πάντων στην, ε, σε Ευρωπαϊκές Τράπεζες Δεδομένων. Εγώ δεν συμφωνώ. Πρέπει νομίζω να υπάρχει ένα νομικό υπόβαθρο για τη χρήση των προσωπικών στοιχείων. γιατί είναι χρήσιμα για την αποφυγή κατάχρησης ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ διοκτικών αρχών να προστατέψουμε άτομα από τα ναρκωτικά αλλά και να καταπολεμήσουμε γενικότερα το οργανωμένο έγκλημα που ασχολείται πολύ συχνά με ναρκωτικά προσπάθησα να εξισορροπήσω την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τη μία με την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος από την άλλη. Το θέμα είναι ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εγώ κατέθεσα την τροπολογία 38 που τα ευθυγραμμίζει όλα με την οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να μπορούμε να ανοιχνεύουμε τα εγκλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να έχουν το δικαίωμα να δίνουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όπως προβλέπει ο κανονισμός. Όλα δηλαδή να γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχει και το θέμα της αποθήκευσης, δύο χρόνια, τρία χρόνια. προτείνω να συναντηθούν οι σκιώδεις αυτή την εβδομάδα ήδη και να αποφασίσουμε αν θα είναι δύο ή τρία χρόνια η κατακράτηση ή η αποθήκευση. Θα τηρήσω ενήμερους όλους τους συντάκτες των τροπολογιών για την πιθανή εξέβρεση, για την εξέβρεση πιθανών συμβιβαστικών. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε την εισηγήτρια. Υπάρχουν σχόλια σχετικά με την έκθεση. Κύριε Φώσου, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Πύρκρο, ο οποίος δυστυχώς ε, κολλείται. Θα ήθελα να τοποθετηθώ συνολικά για την έκθεση αυτή. Όπως είπατε, 46 τροπολογίες κατατέθηκαν και οι τροπολογίες της εισηγήτριας είχαν να κάνουν συχνά με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό αφορά γενικότερα το θέμα. Από πλευρά του ΕΛΚ αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι οι οκτώ τροπολογίες του κυρίου Τριανταφυλλίδη για τη διαγράφη της προτάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, σύσταση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Δεδομένων. Δεν θεωρούμε ότι είναι σωστή η διαγραφή αυτή. Άρα, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για την ε, βάση δεδομένων θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί σε πολύ πρακτικό επίπεδο και από ό,τι κατάλαβα η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σπούκερ. Είναι θετικό το γεγονός ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τροπολογία 38 γίνεται ένα μικρό άνοιγμα για το οποίο είμαστε πολύ ευγνώμονες και στην 39 ο κ. Τσόλκερ αναφέρει το ίδιο πρόβλημα, το θέμα του κατά πόσον επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου με ναρκωτικές ουσίες και πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών. Για την καταπολέμηση της ε, εγκληματικότητας θεωρούμε λοιπόν ότι ε, είναι καλύτερη αυτή η πρόταση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμό και για να διατηρηθεί πρακτικά εφαρμόσιμη αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί η πρόταση η τροπολογία 40 και στην τροπολογία 14 σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να προβλέπονται εξαιρέσεις γιατί μετά από όταν πρόκειται μάλλον για περίπτωση όπου παρεμποδίζονται έρευνες ε, διοικητικές, ε, δικαστικές, σε ό,τι αφορά δίωξη, δηλαδή εγκληματικών δράσεων. Είναι πολύ θετικό σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσα προβλέπονται για τον οξικό ανιδρυτή. Και έχουν κατατεθεί σχετικές τραπολογίες. Συνολικά, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε καλούς συμβιβασμού και αυτό το διευκόλυνα και η συγγήτρια. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερως λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Φως. Η κυρία Εντφέλτ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να μελετήσω ακόμη όλε τι τροπολογίε. Χαίρομαι που ακούω ότι η συγκήτρια από τι αρχή είναι θετική. Η έκθεση επικεντρώθηκε κυρίω σε θέματα προστασία των δεδομένων και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και την άψη του Ευρωπαϊκού από την προστασία των δεδομένων και τη ομάδα εργασία 29. Έχω δύο γενικά σχόλια. Ω γενικό κανόνα να πω ότι δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη ακόμη ότι η δημιουργία νέων βασών δεδομένων ε, για τα πάντα, για κάθε κίνδυνο ή για οτιδήποτε αρνητικό που συμβαίνει στην κοινωνία θα κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Αλλά τέλος πάντων να αφήσουμε τη γενική συζήτηση για κάποια άλλη φορά. Και επίσης θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί το επιχείρημα της δημόσιας υγείας για να αιτιολογήσει παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ, καθώς προέρχομαι από τις κατοχώρες, καλωσορίζω κάτι τέτοιο μεν. Ταυτόχρονα ξέρω ότι σε άλλες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει όχι, όχι, δεν είμαστε αρμόδιοι στον τομέα της δημόσιας υγείας. Υπάρχει λοιπόν κάποιο οπορτουνισμό εδώ, αλλά είμαι έτοιμη να εξετάσω τροπολογίε από κοινού μαζί σα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόγκς. Γενικά είμαι υπέρ ε, του περιεχομένου της τροπολογίας ε, και αναφέρεται σε αυτό συγκεκριμένος ε, τομείς όπου πρέπει να έχουμε μια μεύρη νομοθεσία. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το προτιμούσα, όπω ξέρετε, θα έπρεπε και πάλι να θεσπιστεί με ad hoc διεθνείς συμφωνίες. Πιστεύω ότι η ουσία τη έκθεση αυτή, όταν τροποποιηθεί, γιατί μα είπε ότι ε, η συγκεντρία του θα δεχόταν τις περισσότερες συμφωνίε, συμφωνίες, ε, θα έβρισκε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τη επιβολή του νόμου και τη προστασία των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, Θεωρώ ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τους σπάνιους τομείς που εγώ θα υποστήριζα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά από μένα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κομισιόν, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ μπορώ να είμαι σύντομος, γιατί Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και για την υποστήριξη που έχει δείξει για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ και τους κοιόδες εισηγητές. Συνολικά, οι τροπολογίες που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την προστασία των δεδομένων είναι φυσικά αποδεκτές, δηλαδή η Κομισιόν δεσμεύεται να εφαρμόσει σωστά αυτού τους κανόνες. Επομένως, αν υπομονούμε να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις για τα θέματα αυτά, για να βελτιώσουμε το κείμενο όπου δει. Επίσης, ευχαριστώ την ε, κυρία Χατς και τον κύριο Φως για τα σχόλια στη σχέση με την κατάργηση της βάσης δεδομένων και για να δράση το σχόλιο της κυρίας Σίντβελτ. Ε, η βάση δεδομένων ε, ουσιαστικά αντικαθιστά υφιστάμενες υποχρεώσεις στην τρέχουσα νομοθεσία και με αυτά ε, και αυτές οι υποχρεώσεις γίνονται σεβαστές ε, στέλνοντας email ή αντίγραφα σε χαρτί. Έτσι λοιπόν ε, μας ενδιαφέρουν αυτές οι πληροφορίες αν θέλουμε να συλλεξούμε τα δεδομένα για τις κατασχέσεις και η δεύτερη κυρία λειτουργία της βάσης δεδομένων θα βοηθήσει τις αρχές ε, να δουν ε, κατά πόσο δρούν νόμιμα οι εμποροί αλλά και οι χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά θα αντικαταστήσουμε εδώ τις επιστολές ή τα email. Υπήρχε και μία τροπολογία του κ. Πάρκερ που θα ήθελα να τονίσω, τροπολογία 39. Εδώ προτείνεται οι πληροφορίες που συλλέγονται να χρησιμοποιούνται μόνο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου στα ναρκωτικά και στις προδρόμες ουσίες. Φυσικά αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε επί τις αρχής, όμως να πω ότι έχουμε μια υποχρέωση, δυνάμει της σύμβασης του ΟΗΕ, να κοινοποιούμε τα στοιχεία σε σχέση με τις ε, κατασχέσεις ε, και τις αποστολές ε, που σταματάμε στο τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ. Όμως ε, φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις πληροφορίες. Μιλάμε για τις ποσότητες των πρόεδρων ουσιών που έχουμε κατασχέσει, που τις έχουμε σταματήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν λοιπόν προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Παρακαλώ, συγγητρία. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους για τα θετικά σχόλια. Για την ομάδα του ΕΛΚ, όπως είπα, σύμφωνα μαζί τους, δεν συμφωνώ με την ε, πρόταση της ΓΚΟΕ να διαγράψουμε κάθε αναφορά στη βάση δεδομένων. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν. Κυρία Ιντφελτ. Συμφωνώ με περισσότερο που σα είπατε. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων και των βάσεων δεδομένων κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα θα κάνουμε και μια συζήτηση με τους κοιόδης πολύ σύντομα, θα εξετάσουμε τα κρεμή ζητήματα και θα δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβασμούς. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Δεν υπάρχουν πολλά ακόμα να πούμε. Η ψηφοφορία στη ΛΕΒΕ έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Απριλίου. Αυτά. Επομένω, πρέπει να περάσουμε στην έδραση των συντονιστών. Αν βρίσκονται εδώ στην αίθουσα, παρακαλούνται να μένουν για την συνεδρία και κλεισμένο των θυρών. Και κατόπιν θα συνεχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΠΕ στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Ε? I see that not, not, not all coordinators are here. So, again, 15 minutes of recess. 15 λεπτά διάλειμμα, έτσι ώστε οι συντονιστές που δεν είναι στην αίθουσα να μπορέσουν να έρθουν. Our schedule for 10:45 can make it to the to the room of the meeting. Thank you.